και τους λόγους για την ε, υιοθέτησή τους, καθώς και τη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τίτλοι θα περιληφθούν στα πρακτικά της παρούσας συνόδου και το τρίμηνο που έχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να στη θέση του θα αρχίσει να τρέχει από αύριο 20 Φεβρουαρίου του 2009. Τα πρακτικά της συνεδρίασης θα υποβληθούν στο